δύσκολη αυτή η δουλειά και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε και έχει άρα ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει εδώ το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω λάβει ένα ψήφισμα, μια, ένα ψηφίσματος για το κλείσιμο της συζήτησης. Αύριο στις 11.30 θα γίνει η ψηφοφορία. Έχει λήξει λοιπόν η συζήτηση. Μια σύντομη ανακοίνωση για την πρόταση διορισμού βουλευτών στην Ειδική Επιτροπή για το Οργανωμένο ε, Έγκλημα, την ε, ε, λεύκανση χρημάτων κτλ. Όλα αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και η προθεσμία για τι τροπολογίε σε αυτή την πρόταση θα είναι αύριο. Και θα ψηφιστεί αύριο η πρόταση για τη σύνθεση αυτή τη Επιτροπή. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η δήλωση του Συμβουλίου